Καλημέρα, συνάδελφοι. Η συνεδρίασή μας σήμερα είναι από τις 9.30 μέχρι τις 11.30 και μετά έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών μέχρι τις 12.30 για την έγκριση της ημερήσιας διάταξης έχουμε κάποιες αλλαγές. Το σημείο 4 για το Eurodac έχει αναβληθεί. Επίσης, στις 11 και 10 έχουμε δύο ψηφοφορίες. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε εγκρίθηκε. Για τα γλωσσικά, δυστυχώ ε, κροατικά, λετωνικά και γαλλικά δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν δανέζικα το απόγευμα. Περνάμε τώρα το άρθρο 205 έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Έχουμε κάποιες επιπρόσθετες ημερομηνίες συνεδρίασης 11 Απριλίου 9 με 12.30 και 27 Απριλίου από 2 με 5.30 το απόγευμα. Εγκρίνεται, ναι, ωραία. Τρίτον, Ενημέρωση για τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δευτέρα 3 Απριλίου 16 κράτη-μέλη ειδοποίησαν Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν σύμφωνα με το άρθρο 86 την επιθυμία να υπάρξει ενηχημένη συνεργασία για τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα θα οριστικοποιηθεί το κείμενο και θα πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο κανονισμού από το Κοινοβούλιο και αφορά 16 κράτη-μέλη. Σημείο 4 για την ε, λεγόμενη Επιτροπή χωρίς χαρτιά. Ίσως θυμάστε πως στην αρχή της αιτίας ε, ε, είπαμε για μια σταδιακή προσέγγιση για να μην εκτυπώνουμε έγγραφα. Σας ενημερώσαμε τότε για την εφαρμογή στο διαδίκτυο, την e-meeting, όπου υπάρχουν όλα τα έγγραφα. Ίσως λοιπόν να προσέξατε ότι σταμάτησε η διανομή των εγγράφων ε, και μπορείτε να τα ζητάτε από τους κλητήρες γιατί σχεδόν όλα αυτά παραμένουν αχρίαστα. Οπότε περνάμε τώρα στην τελική φάση και σταματάει η εκτύπωση των εγγράφων. Οπότε από σήμερα θα τυπώνεται μόνο η μερίσια διάταξη. Οπότε οι βουλευτές που δεν χρησιμοποιούν ακόμα την εφαρμογή e-meeting παρακαλώ να ενημερωθούν και να κατεβάζουν τα σχετικά έγγραφα. Τέλος, να επαναλάβω. Ναι αν συμφωνείτε όλοι πείτε μου το 5 είναι οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να έχετε την κάρτα στις 11 και 10 τέλος έγκριση πρακτικών 27 με 28 Φεβρουαρίου και 23-24 Μαΐου και 23 και 24 Μαρτίου, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνονται. Το σημείο 4 αναβλήθηκε και περνάμε στο σημείο 5. Έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή και την εκφόρηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό του 2013 για πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών σύμφωνα με τα άρθρα 14.1 και 18.2 ε, ε, του κανονισμού που εγκρίθηκε πέρσι τον Φεβρουάριο, οπότε θα δώσω τον λόγο στην Κομισιόν για μια σύντομη παρουσίαση και μετά σε κάποιον βουλευτή, αν επιθυμεί. Ο κύριος Ντάς από την Κομισιόν για 5 λεπτά. Να έχετε τον λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που βρήκατε κάποιο χρόνο για αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πιστεύουμε ότι η καταπολέμηση της ε, απειλής ε, των εκρηκτικών που κατασκευάζονται στο σπίτι παραμένει ε, ουσιαστικά μία από τι κύριε προτεραιότητε για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Ακόμη και αν οι πιο πρόσφατε επιθέσει στην Ευρώπη έγιναν με άλλα μέσα, τα εκρηκτικά που κατασκευάζονται στο σπίτι, ε, μαζί με τα συμβατικά πυροβόλα όπλα, είναι τα προτιμόμενα από τους ε, τρομοκράτες γιατί είναι πολύ αποτελεσματικά και διαθέσιμα και είδαμε ουσιαστικά την καταστροφική επίδραση και στην Αίγυπτο και στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι. Η προπαγάνδα στο ίντερνετ δίνει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση σε πιθανούς τρομοκράτες, σε οδηγίες για την κατασκευή ε, βομβών και στο Καλυφάτο είδαμε μια μεταφορά γνώσης ε, σε ό,τι αφορά τους ευθοσχέδιους εκρηκτικούς ε, μηχανισμούς και Υπάρχει με την επιστροφή των μαχητών στην Ευρώπη κάποιος φόβος ε, ότι θα μπει αυτή η γνώση και στην Ένωση. Έχουμε λοιπόν ε, πολύ καλούς λόγους ε, να συνεχίσουμε και να ενισχύουμε τη δουλειά της προστασίας μας κατά των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και βλέπουμε ότι χρειάζεται σε αυτό το τομέα μια κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δυσκολεύσουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών σε αυτά τα χημικά. Και γι' αυτό το 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέτησαν τον κανονισμό 98 κάθετος 2013 σε ό,τι αφορά την εμπορία και τη χρήση των πρόδρομων ε, ουσιών, των εκρηκτικών, ε, για να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα των χημικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τέτοιων εκρηκτικών ε, και επίσης να μπορούμε να παρακολουθούμε και τις ύποπτε συναλλαγές. Στα τέλη του Φεβρουαρίου η Κομισιόν θέτησε μία έκθεση για τον κανονισμό αυτό, που συνδυάζει δύο σκοπού. Καταρχήν την υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή του κανονισμού και δεύτερον για το πώς εκτελεί η Κομισιόν ε, τις εκτελεστικές πράξεις. Ε, επίσης, ε, η συλλογική μας εμπειρία πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μικρή και δεν μπορούμε να εξαγάγουμε ακόμα τελικά συμπεράσματα. Η Κομισιόν σκοπεύει με την εκθεσία αυτή να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει γίνει προς ε, το να κάνουμε ασφαλείς ε, ε, αυτές τις πρόδρομες ουσίες και δεύτερον να δούμε τι αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αλυσίδια εφοδιασμού και να ενισχύσουμε τις μελλοντικές προσπάθειες αλλά και τελικά να διευκολύνουμε την άσκηση κατεξουσιοδότηση πράξεων. Πιστεύουμε ότι ο κανονισμός πράγματι συνεισφέρει στη μείωση των απειλών που τίθεται από τέτοιους αυτοσχέδιους μηχανισμούς ε, στην Ευρώπη. Καταρχήν έχει μειωθεί ο απόλυτος αριθμός ε, των πρόδρομων χημικών ουσιών που είναι διαθέσιμες στην αγορά της Ευρώπης. Φαίνεται ότι βλέπουμε μία μετακίνηση προς εναλλακτικές ουσίες που είναι λιγότερο επικίνδυνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς, αλλά όχι ε, για τους ίδιους σκοπούς στο νοικοκυριό δηλαδή, αλλά όχι για την ε, παρασκευή χημικών ε, για την παρασκευή βομβών. Επίσης, παρακολουθούμε διάφορες ύποπτες περιπτώσεις. Έχουν αναφερθεί διάφορες ύποπτες συναλλαγές εξαφανίσεις και κλοπές αυτών των χημικών. Η έκθεση επίσης τονίζει ότι υπάρχουν κάποιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για τα κράτη-μέλη. Οι κύριες προκλήσεις ε, είναι να απευθυνθούν στην πολύ μεγάλη λύση διαφοδιασμού. Μιλάμε ουσιαστικά για προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο νοικοκυριά και επίσης ε, να αντιμετωπίσουμε και διάφορες ε, άλλες μορφές πώλησης, παραδείγματος χάρη μέσω του διαδικτύου. Οι κύριε προκλήσει για την αλυσίδα εφοδιασμού είναι να εντοπίσουν όλα τα ενδιαφερόμενα προϊόντα, να αξιολογήσουν ε, αν είναι επαγγελματίε ή χρήστε ή το γενικό κοινό, γιατί γίνεται μια διάκριση από τον κανονισμό και να δουν αν είναι οι συναλλαγές ύποπτε. Ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ είναι για το αν ε, το πεδίο του περιορισμού θα πρέπει να καλύψει και τους επαγγελματίες χρήστες των ουσιών και όχι μόνο τα μέλη του γενικού κοινού. Πέρα από την καλή δουλειά που έχει γίνει, με τον κανονισμό είδαμε και παραδείγματα όπου οι τρομοκράτες συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τις πρόδρομες ε, χημικές ουσίες και η Κομισιόν σκοπεύει να αναθεωρήσει τον κανονισμό προκειμένου να αντιμετωπίσει και αυτές τις προκλήσεις και να ενδυναμώσει το σύστημα γενικώ στο μέλλον. Σκεφτόμαστε ή να έχουμε πιο ισχυρού περιορισμούς και ελέγχους ε, σε κάποιες νέες ουσίες, ή ήδη κατεχωρημένες ουσίες. Επίσης προτείνουμε να αποσαφηνίσουμε και να εναρμονίσουμε κάποιες από τις διατάξεις, κυρίως όταν βοηθά αυτό την αλυσίδα εφοδιασμού να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της πιο αποτελεσματικά και ευρύτερα θα αξιολογήσουμε τα το κόστος και τα ωφέλη πρόσθετων μέτρων, είτε κανονιστικών είτε μη κανονιστικών, που θα αυξήσουν την ικανότητα όλων των ενεχόμενων φορέων. Και τέλος, στην έκθεση σημειώνουμε ότι η Κομισιόν χρησιμοποίησε τις κατεξουσιοδότηση αρμοδιότητές της το 2016 για τρεις ουσίες στο παράρτημα 2 η σκόνη αλουμινία, το νητρόδες μαγνήσιο και σκόνη μαγνησίου. Θέλω να ποτίσω φοροτιμή ε, στο έργο που έγινε στη μόνιμη επιτροπή για τι πρόδρομε ουσίε, όπου βλέπουμε μια πολύ θετική δυναμική και μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τη Κομισιόν και μια πολύ θετική δυναμική στον τομέα αυτό. Η Κομισιόν λοιπόν ε, παραμένει απόλυτα δεσμευμένη για την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού και αξιολογούμε προσεκτικά την ανάγκη και τον πιθανό αντίκτυπο νέων περαιτέρω μέτρων σε αυτό το τομέα. Επίσης, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και με τη δική σας επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω αν κάποιοι βουλευτές θέλουν το λόγο. Κυρία Σίπελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ για να καταλάβω καλύτερα τι συμβαίνει. Δεν θα σκέσω κριτική. Αναφέρεται ότι έχουμε πολλές αναφορές για ύποπτες συναλλαγές. Αυξάνεται ο αριθμός επειδή αυξάνεται και η ευαισθητοποίηση στον τομέα αυτό. Και αυτό μας οδηγεί σε σαφή αποτελέσματα ότι υπάρχουν προβληματικές συναλλαγές οι περισσότερες από αυτές τις συναλλαγές είναι νόμιμες τελικά ή οδηγούν σε κάποια ποινική έρευνα και σε σχετικά αποτελέσματα. Η έκθεση αναφέρεται στην ε, κατεξιοδότηση αρμοδιοτήτων, στην αρμοδιοτήτων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη. η Κάποιος άλλος πριν απαντήσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρικίτη ο πρόσωπος της Κομισιόν, κύριο Τάσο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Βλέπουμε αρκετά αποτελέσματα και μερικές φορές ε, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τη σχέση μεταξύ των διαφορών φορέων των διαφοροπαραγόντων. παραγόντων. βλέπουμε ότι μειώνεται ο αριθμός των πρόδρομων ουσιών και αυτό εν με στο ότι οι πολλοί οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τους περιορισμούς και εν μέρη επειδή εκούσια κάποιοι παρασκευαστές σταμάτησαν την παραγωγή αυτών των ουσιών ή κάποιοι οικονομικοί φορείς σταμάτησαν να πουλάνε αυτές τις πρόδρομες ουσίες των εκρηκτικών. Και η αλυσίδα εφοδιασμού δεν μας ε, έφερε σημαντικές ε, οικονομικές απώλειες ή ε, διαταραχές ως αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ότι υπάρχει λιγότερη γοροπολισία των ουσιών. Επίσης ε, είδαμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των αναφερόμενων υπό των συναλλαγών ε, και της αναφοράς κλοπών ή εξαφανίσεων. Αυτό οφείλεται και στο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μεταξύ των οικονομικών φορέων, γίνονται πιο προσεκτικοί, επαγρυπνούν, για να το πούμε πιο απλά, και επίσης επειδή υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των διοκτικών αρχών και μεγαλύτερη πίεση επί των οικονομικών φορέων. Κάποια κράτη-μέλη σε μια βάση ad hoc ε, αντίλαξαν πληροφορίες ε, για τις ε, εκθέσεις και για τις άδειες που ήταν αντικείμενο άρνησης, όμως νομίζω ότι είναι κάπως σκόρπιες αυτές οι πληροφορίες. Είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Θα έχουμε νομίζω ξεκαθαρή εικόνα σε λίγα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα την εκτέλεση των εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων. Έχουμε χρησιμοποιήσει τις κατεξουσιοδότηση αρμοδιότητες, αυτές τις τρεις ουσίες που σας ανέφερα στο παράρτημα 2, τις προσθέσαμε εκεί, δηλαδή υπόκεινται σε έλεγχο. Αυτό έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο, βάση πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ζήτηση προήλθε από τη μόνιμη επιτροπή για τι πρόδρομες ουσίε. Δηλαδή τα ίδια τα κράτη-μέλη πίστευαν ότι αυτές οι τρει ουσίε θα πρέπει να προσταθούν στον κατάλογο. Οι προτάσει κοινοποιήθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέσω τη κανονική διαδικασία και δεν λάβαμε αντιρρήσει ή σχόλια. Υιοθετήθηκαν επομένω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε επικεφαλή ε, της ε, Μονάδας ε, για την Καταπολέμηση τη Δημοκρατίας και της ρίζου πεστικοποίηση. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια και ερωτήσει. ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή για την παρουσίαση. Ευχαριστώ και την Μπριγκίτ για αυτή τη σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Α περάσουμε τώρα στα σημεία 6 και 7 για την επιστροφή, συγγνώμη, πολιτική επιστροφών. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 2 ε, Μαρτίου εφέτησε σύσταση για το πώ θα καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την πολιτική επιστροφών ε, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, παρέχοντα έτσι καθοδήγηση προ ε, τα κράτη-μέλη για το πώς οι διατάξεις τη οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζονται. Και στις 3 Φεβρουαρίου λοιπόν υπήρξε ε, αυτή η κίνηση και η σύσταση συνδέεται με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανανεωμένο σχέδιο δράσης για τις επιστροφές ε, με μια ειδική έμφαση ε, στις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνονται. Θα δώσουμε το λόγο το, τώρα στον κύριο Τουντοράς από τη Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων, επικεφαλής της ε, Μονάδας για την Παράτητη Μετανάστευση και την Πολιτική Επιστροφών. Είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, εξέτοιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θεωρεί την διαχείριση της μετανάστευσης ως μία σειρά δράσεων και ενεργειών ε, που βέβαια θα πρέπει και να προστατεύουμε τα δικαιώματα των μεμονωμένων ατόμων αλλά και ε, να ρυθμίζουμε τη μετανάστευση πάντα με συγκεκριμένε και υπεύθυνε δράσει. Η πολιτική επιστροφών θα πρέπει να βασίζεται και στι εσωτερικέ δράσει σε επίπεδο 100 μελών, αλλά και στη συνεργασία με τρίτε χώρε ε, για να διασφαλίσουμε την επανεσδοχή τους. Το 2015 η Κομισιόν υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης για τις επιστροφές. Συμπεριλάμβανε 40 πολύ καλέ ε, ενέργειε, πολλέ από τι οποίε έχουν ήδη υιοθετηθεί. Όμω αυτό το σχέδιο δράση υιοθετήθηκε και υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό πριν από τη μεταναστευτική κρίση. Γι' αυτό, αν δούμε τα στοιχεία σήμερα, θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να επικαιροποιηθεί το σχέδιο δράση αυτό. έχουμε μείνει περίπου στο 35% με 40% στο ποσοστό επιστροφών τα τελευταία χρόνια. Αν αφαιρέσουμε τις επανεισδοχές στα Δυτικά Βαλκάνια ή στις χώρες της Ανατολικής Τερικής Σχέσης, με τις οποίες έχουμε πολύ καλές ε, συμφωνίες που λειτουργούν πολύ καλά για την επανεισδοχή, τότε αυτό το ποσοστό ε, πέφτει κάτω το 30%. Από την άλλη, φτάνουμε στη στιγμή όπου οι πάνω από, το, από ένα εκατομμύριο τούτε άσυλο που έχουν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ε, θα λάβουν ε, οριστική απόφαση και αρκετοί από αυτούς ε, θα λάβουν αρνητική απάντηση. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και εμείς και τα κρατημέλη μας για αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι και ο σκοπό του νέου αναθεωρημένου σχεδίου δράση και τη δέσμη που υιοθετήσαμε. Το σχέδιο δράση δηλαδή και οι συστάσει λαμβάνουν υπόψη αυτές ε, τις ε, συγκυρίες και το χαρακτήρα του κατεπήγοντος που προκύπτει στα κράτη-μέλη και εξετάζουμε πώς τα κράτη-μέλη αξιοποιούν το νομοθετικό, επιχειρησιακό και ε, οικονομικό πλαίσιο εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους. Τι συμπεριλαμβάνει το αναθεωρημένο σχέδιο δράση επιχειρεί να δούμε πώς τα εθνικά συστήματα και οι διαδικασίες επιστροφής μπορούν να καταστούν πιο αποτελεσματικά, ε, αξιοποιώντας καλύτερα την οδηγία περί επιστροφών. Γι' αυτό στη δέσμη υπάρχει και σύσταση που εξετάζει σε βάθος πώς τα κράτη-μέλη έχουν υλοποιήσει την οδηγία μέχρι σήμερα και πώς την έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο. Και θα φτάσω στη σύσταση που είναι ξεχωριστό έγγραφο. Δεύτερον, Εξετάσαμε πω στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι διαδικασίε ασύλου μπορούν καλύτερα να συνδεθούν, ε, να διασυνδεθούν με την πολιτική επιστροφών για να υπάρχει συνέπεια, συνοχή και συνέργειε σε εθνικό επίπεδο για την ε, εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Τρίτον, το σχέδιο δράσης μιλά για περαιτέρω βελτίωση τη ανταλλαγή ε, πληροφοριών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μεταξύ κρατών μελών και με, με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έχουμε κάποια συστήματα πληροφορικής αυτή τη στιγμή που είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές. Εξετάσαμε την πρόσβαση ε, των ε, αρχών ε, στις βάσεις αυτές και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την πρόσβαση. Τέταρτον, βελτίωση της ανταλλαγής των πρακτικών για να διασφαλίσουμε ε, συνέπεια και συνοχή σε ό,τι φορά την πολιτική επιστροφών. Μιλούμε επίσης για εναρμόνιση των ε, ε, πακέτων εθελούσιας επιστροφής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τρίτες χώρες που κάνουν forum shopping για τα καλύτερα πακέτα επανεισδοχής. Θέλουμε να βελτιώσουμε επίση τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδίω σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή. Θέλουμε να αυξήσουμε το προσωπικό και να θεσπίσουμε και έναν ε, μηχανισμό χρηματοδότηση των επιστροφών μέχρι τον Ιούνιο. Περιμένουμε επίση από αυτόν τον οργανισμό να αυξήσει ε, τι ε, ε, των τρίτων, για τι τρίτε χώρε ό,τι αφορά την επιστροφή μέχρι τον Οκτώβριο. Θέλουμε αυξημένη οικονομική στήριξη μέχρι και 200 εκατομμύρια ε, ευρώ για τις εθνικές προσπάθειες επιστροφών. Και το σχέδιο δράση εξετάζει τι προκλήσει τη επανεισδοχή, γιατί οι ενέργειε σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει κάπω να εξισορροπούνται μέσω τη αποτελεσματική συνεργασία με τρίτε χώρε. Ανέφερε και τη σύσταση μαζί στη δέσμη. Βασίζεται στην οδηγία περί επιστροφών και εξετάζει πολύ ρεαλιστικά με βάση και την αξιολόγηση Σέγγεν που έγινε στα κράτη-μέλη τα τελευταία δύο χρόνια για να δούμε πώς ακριβώς μπορούν καλύτερα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τους κανόνες ε, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί επιστροφών. Δεν προβλέπονται νέες υποχρεώσεις παραμένουμε εντός των ορίων που προβλέπονται ε, στην οδηγία. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι μια ενιαία σύσταση για όλους με τον ίδιο ομοιόμορφο τρόπο από όλα τα κρατημέλη. Υπάρχουν ε, ενδέχεται μάλλον ορισμένες συστάσεις να είναι πιο συναφείς και σημαντικές για κάποια ε, κρατημέλη από ότι για άλλα, ανάλογα με την κατάσταση. Όμως θέλουμε όλα τα κρατημέλη να εξετάσουν ε, με κριτική ματιά ε, αυτές τις συστάσεις για να δουν τι πραγματικά τους χρειάζεται. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και αρχών ούτω ώστε οι δεξιότητε και η προγραμμοσύνη που χρειάζονται να είναι διαθέσιμα για να έρονται τα εμπόδια ε, που υπάρχουν για την επιστροφή. Εξετάζουμε διαδικαστικές και επιχειρησιακές ε, αδυναμίες στα κράτη-μέλη και τις αρχές. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις Και θέλουμε να εντοπίζουμε αυτέ τι καταχρήσει όταν γίνονται μόνο και μόνο για να καθυστερήσουν το αναπόφευκτο, δηλαδή την τελική επιστροφή. Ε, θέλουμε να κάνουμε καλή, σωστή χρήση τη απαγόρευση εισόδου θέλουμε να θεσπίσουμε ένα πρόγραμμα εθελούσες επιστροφής μέχρι τον Ιούνιο 2017 και να διασφαλίσουμε μια καλή ε, ανταλλαγή πληροφοριών. Δύο σημεία τώρα τα οποία ε, έτυχαν ιδιαίτερο ενδιαφέροντος από την κοινωνία των πολιτών και έχουν συζητηθεί επί μακρόν τις τελευταίες εβδομάδες ήταν οι συστάσεις σχετικά με την κράτηση και τους ε, ανηλίκους. Για την κράτηση η σύσταση ε, προσφέρει πιο σαφείς ε, προβλέψεις για το πώς θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται η οδηγία για να εξοποιείται σωστά το πλαίσιο που προβλέπει η οδηγία για την κράτηση. Δεν κάνει λόγο για κράτηση ως αυτοσκοπό. Απλώς ε, και πάλι περιμένουμε τα κράτη-μέλη ότι θα κάνουν μια πιο έξυπνη χρήση της ε, πραγματικότητας και της νομοθεσίας ε, για να ε, βελτιώνει τα συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία και υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής, τότε η κράτηση θα πρέπει, μπορεί και θα πρέπει να αξιοποιείται, ούτως ώστε να καθίστανται δυνατές αυτές οι επανεισδοχές. Όταν δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία επανεισδοχής, βέβαια δεν περιμένουμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν αδιακρίτω κράτηση με σκοπό την επιστροφή όταν είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επανεισδοχή. Σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους, είτε είναι ασυνόδευτοι είτε όχι, το πρώτο που επισημαίνει η σύσταση είναι η διασάφηση του ε, νομικού καθεστώτος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο σε εθνικό επίπεδο. Γιατί το ασαφές νομικό καθεστώς για τους ανηλίκους ενδέχεται να τους ε, οθήσει προς ε, τη φέα ζώνη και προς προβληματικές καταστάσεις. Δεύτερον, η σύσταση θεωρεί ότι ως ε, μέρος ε, της πλήρους αξιολόγησης κάποιες φορές η επιστροφή του ανηλίκου στην ε, οικογένειά του στη χώρα προέλευσης ενδέχεται να είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου. Και αυτό πάλι όχι τυφλά και αδιάκριτα, αλλά ως μέρος μιας πολυσχηδούς αξιολόγησης. Όμω πάντα η επιστροφή στην οικογένεια θα πρέπει να είναι τμήμα μέσα στο φάσμα των ενεργειών που έχει στη διάθεσή του το κράτος μέλο. Λοιπόν, έχουμε ένα φιλόδοξο πακέτο λοιπόν ε, που απαιτεί επένδυση σε ανθρώπινους, οικονομικούς και πολιτικούς ε, πόρους και είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Θα υποβάλουμε έκθεση για την πρόοδο που θα σημειωθεί για το αναθεωρημένο, ε, σχέδιο δράσης μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς είναι σημαντικό και ευαίσθητο το θέμα. Περνάμε τώρα στους ομιλητές. Ξεκινάμε την κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για το ότι ήταν τόσο λεπτομερής. Να πω ξεκάθαρα ότι Υπάρχει μία πτυχή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης όπου ακόμα απέχουμε πολύ από το να εφαρμόζουμε κάτι είναι οι επιστροφές. Αν δούμε τους αριθμούς ατόμων που επιστρέφονται είναι εξαιρετικά χαμηλοί λόγω των παραγόντων που μόλις αναφέρθηκαν και βεβαίως πρέπει να τονίσουμε την σημασία όλα τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται για να υπάρχει ένα σύστημα ενιαίο σε ολόκληρη την Ένωση. Και ακριβώ το ότι διαλέγουν κάποιοι κάποια κράτη-μέλη λόγω των πακέτων εθελοντικής επιστροφής προσφέρονται είναι πολύ σημαντικό. Να αναφερθώ στη χώρα μου, όπου υπήρχαν ε, επιτυχημένα προγράμματα εθελοντικών επιστροφών που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει για να επιστραφούν τα άτομα σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Αλλά και εδώ πέρα επίσης οι λέξεις ε, δυνατό και πρακτικό που ανέφερε η Κομισιόν έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί εάν η επανεισδοχή δεν είναι δυνατή, αν ένα κράτος μέλος δεν έχει διμερείς διευθετήσεις με μια τρίτη χώρα, τότε ποιος είναι ο ρόλος της ε, Κομισιόν όπως ζητάει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπέρασματά του. Και κάθε τρεις-τέσσερις μήνες ε, ακούμε ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα αρκετά για την υπηρεσία ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής και εδώ πέρα βεβαίως αναμένουμε να δοθεί περισσότερη έμφαση γιατί έχουμε προθεσμίες ε, και περιμένουμε, περνάνε οι μήνες και βλέπουμε πως τα όσα συμφωνήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο δεν έχουν εφαρμοστεί. Για τους ανήλικους, τέλος, η διευκρίνηση του νομικού καθεστώτος έχει μεγάλη σημασία. Γνωρίζουμε τις διάφορες μεθόδους ε, που χρησιμοποιούνται σε διάφορα κράτη-μέλη. Είναι σαφές πως αυτή τη στιγμή υπάρχει κατάχρηση πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι αγνοούνται, ε, αποτελούν αντικείμενο αδικημάτων και πρέπει να συνεργαστεί η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ. Μπίργκιτ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές. Μπορεί να αρέσει σε κάποιους ή όχι, αλλά γεγονός είναι πως το στοιχείο των επιστροφών είναι μέρος του συστήματος ασύλου. Όσοι λοιπόν ετούνται άσυλο αλλά τελικά απορρίπτονται πρέπει να επιστραφούν ε, σε έναν ιδεώδη κόσμο στην χώρα προέλευσής τους. Οπότε το πρώτο ερώτημα, ναι, συμφωνώ όταν μιλάμε για επιστροφές ε, χρειάζονται σαφείς κανόνες για το πώς θα γίνονται, για να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και να γίνεται με τρόπο αποδεκτό. Το δεύτερο ερώτημα λοιπόν είναι επιστρέφουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους ε, στις χώρες προέλευσης ή σκεφτόμαστε να τους επιστρέψουμε και σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Και στο μέτρο αυτό γιατί θα πρέπει να δεχτεί οποιαδήποτε τρίτη χώρα ανθρώπους που δεν είναι υπηκόου ε, Μπορεί να τους πληρώνουμε, αλλά ανησυχώ για το πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε. Αν δεν είναι ζήτημα χρημάτων που δίνουμε σε τρίτες χώρες, αλλά εμείς ε, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ασχοληθούμε με αυτούς και ζητάμε από άλλες τρίτες χώρες να το κάνουμε. Οπότε εγώ θα ήθελα να επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι ή δυνατόν στις χώρες προέλευσης. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η συνάδελφος κυρία Μέτσολα ανέφερε και γεγονός είναι πως έχουμε κάποιες διμερείς συμφωνίες επιστροφών. Αλλά δεν θα έπρεπε να έχουμε ε, ευρωπαϊκές ε, συμφωνίες επανεισδοχής. Γιατί ε, δεν νομίζω ότι βοηθάει μία χώρα να έχει συμφωνία επανεισδοχής με μια χώρα ε, προέλευσης. Οπότε μια χώρα έχει την ευκαιρία να στείλει ε, κόσμο στην ε, χώρα προέλευσης, αλλά οι άλλες 27 να μην έχουν. Τι λέμε λοιπόν όταν μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκές συμφωνίες επιστροφών και επανεισδοχής και όχι 27 ή 28 διμερείς συμφωνίες. Εάν θέλουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, βεβαίω θα θέλαμε να προστατεύσουμε τον κόσμο ο οποίος φεύγει για να γλιτώσει από βασανιστήρια, από όλεμο κτλ. Αλλά όχι βεβαίως όσους είναι α, ε, φτωχοί. Θεωρώ λοιπόν πως οι διαδικασίες ασύλου θα πρέπει να είναι νομικά στερεές αλλά και κάπως πιο γρήγορες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόσμο για ένα χρόνο ή και παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο τότε να αποφασίσουμε ότι πρέπει να επιστρέψουν. Κανείς δεν κατανοεί κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να προστατεύσουμε μόνο όσους έχουν δικαίωμα σε άσυλο, τότε πρέπει να ε, δούμε το ζήτημα. Και το ερώτημά μου είναι, έχετε κάποια πληροφορία ότι τα κράτη-μέλη μας εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι θα έχουν θα επιταχύνουν την διαδικασία αυτήν. Τώρα το θέμα είναι η συνεργασία με τρίτες χώρες. ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα εξετάσουμε. Μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά μέτρα γιατί η κατάσταση διαφέρει αναχώρα χώρα προέλευσης. Μιλάμε μόνο για περιοριστικά μέτρα για τις χώρες αυτές. Μιλάμε για αλλαγή της εξωτερικής μας πολιτικής μεταξύ των οποίων η ενέργεια, το εμπόριο, η αλληλεία κτλ. Ποια είναι η στρατηγική μας εδώ και βλέπετε κάποια πρόοδο στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ κύριος Κώστερ. Ήθελα να τονίσω ότι σε σχέση με απορριφθήσεις αιτήσει ασύλου το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση του κράτους και της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να είναι αυτό ένας προσανατολισμός μας και όταν μιλάμε για άτομα των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί. Και έχω αμφιβολίες για το αν αυτό τηρείται πάντα. Και θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι τι πρόθεση έχουμε, ε, πώς θα συλλαμβάνουμε άτομα στα σύνορα όταν ε, πώς θα συμβαστεί αυτό δηλαδή ε, με την γενική αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας. Κάτι το οποίο πρέπει και να ισχύει και για άτομα τα οποία εμφανίζονται στα εξωτερικά σύνορα ως πρόσφυγες ή μετανάστες. Δεύτερον, τι κάνουμε με τους ανηλίκους. Η αρχή πρέπει να είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατεύεται το παιδί και εδώ πέρα αναρωτιέμαι ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλυφθούν για να διασφαλίσουμε την ευημερία του παιδιού και να υπάρξει ενίσχυση της επανένωσης οικογένειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Διάς Δεμέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό το σημείο βασίζεται στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας περί επιστροφών και στην ανακοίνωση της Κομισιόν για πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Αυτό είναι το σημείο εφετηρίας. Όμως, εγώ θέλω να επενθυμίσω ότι η οδηγία επιστροφών ήταν μια κεντρική συζήτηση στη θητεία 2004-2009. Όπως θα θυμούνται και ο Κάρλος και άλλοι, η οδηγία αυτή προχώρησε λόγω της υποστήριξης ε, των δύο μεγαλύτερων ομάδων του Κοινοβουλίου, την υπερψήφισε το ΕΛΚ, το οποίο τότε συμπεριλάμβανε και τους ε, Βρετανούς συντηρητικούς ε, και την ψήφισε και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με την εξαίρεση δύο Ισπανών, ο ένας ήταν ο κύριος Βιόλς και ο άλλος ήταν ο κύριος Μπορέλ. Αυτό ήταν το σημείο Επίσης είναι αλήθεια ότι ήταν μια πολεμική οδηγία. Ένα σημαντικό ζήτημα που θέλω να θέσω σε ερώτηση είναι πόσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεταφέρει στο εσωτερικό τους δίκαιο την οδηγία, πόσες χώρες την έχουν εφαρμόσει και πόσες όχι, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδος, ιδίως για την Ελλάδα, λόγω της ε, νησιωτικής ε, της κατάστασης. Θέλω να πω και το εξή. Αν, θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, είπε ο μιλητής ότι υπάρχει πίεση από την κοινωνία των ε, πολιτών σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους και το θέμα της κράτησης. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να καλέσουμε εδώ τους γλωσσομαθείς νομικούς, γιατί εγώ όπως θυμάμαι στην οδηγία επιστροφών δεν ε, ε, αναφέρεται καθόλου η λέξη κράτηση, detention, φυλάκιση, αλλά αναφέρεται η διοικητική κράτηση, όχι η ποινική φυλάκιση. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό η Επιτροπή και το Συμβούλιο να ξεκαθαρίσουν το θέμα της χρήσης των ενιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές όταν αξιολογούμε και θέτουμε σε εφαρμογή την πολιτική επιστροφών. Γιατί στην οδηγία, από θυμάμαι, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε φυλάκιση, detention. Και εδώ μιλήσαμε για detention και για την μεταχείριση σε σχέση με την φυλάκιση. Θυμάμαι ότι προσπαθούσαμε το 2007 να δώσουμε νομική ασφάλεια σε ό,τι αφορά την περίοδο της διοικητικής κράτησης και βάλαμε το όριο σε 18 μήνες, αν ε, θυμάμαι καλά. Μου γνέφει καταφατικά και ο Κάρλος που σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, εγώ ήθελα να ξέρω αν όντως μετά από τους 18 μήνες διοικητικής κράτησης και της νομικής δυνατότητας ε, αυτός ο πολίτης ε, του οποίου δεν έχει προσδιοριστεί η υπηκότητα ή που δεν έχει γίνει δεκτός, ε, δεκτή επιστροφή του βάση διμερούς ή άλλη συμφωνίας, τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς. Και αν η ανακοίνωση της Κομισιόν ε, για την αποτελεσματική εφαρμογή των επιστροπών λαμβάνει υπόψη αυτές τις τυχές. Φυσικά εκφράζω και την ανησυχία μου για την κατάσταση των ανηλίκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δίας Δεμέρα. Είναι πολύ χρήσιμο που μας υπενθυμίζετε την οδηγία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την πολιτική της φυλάκησης αλλά μας είπατε ότι ο όρος detention δεν αναφέρεται στην οδηγία, όμως το εγχειρίδιο της Κομισιόν αναφέρει τον όρο detention και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η φυλάκηση είναι αρμοδιότητα των ε, κρατών μελών. Όμως ε, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτό το θέμα και να ρωτήσω την Κομισιόν. Ανησύχηση κοινωνία των πολιτών, ε, είπατε, ισχύει τόσο είπε ο κ. Δίας Δεμέρα για το πώς περιλαμβάνεται στην οδηγία. Όμως θέλω να ρωτήσω, το εγχειρίδιο της Κομισιόν λέει ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματικά. Ποια είναι η άποψη της Κομισιόν σε σχέση με το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιούν ε, ε, αυτή τη σε πιο συστηματικά όπως είπε υπονοεί η Κομισιόν στο εγχειριδιό τη. Τι έχετε να πείτε σε σχέση με το όσο είπε και ο κύριο Δεμέρε ότι δεν υπάρχει όρος στην οδηγία. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, κύριο Ράντεφ. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στη Στοκχόλμη τις προηγούμενες μέρες ε, και στο Βερολίνο πέρσι μας ε, έδειξαν ότι πρέπει να έχουμε ταχείς διαδικασίες για την επιστροφή των μεταναστών που δεν πληρούν τα κριτήρια διεθνούς προστασίας πράγματι οι διαδικασίες συναντούν πρακτικές δυσκολίες. Αλλά αν θα πρέπει τελικά να βελτιώσουμε την προστασία όλων όσων έχουν δικαίωμα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πρέπει να συνεργαζόμαστε καλά με τις τρίτες χώρες και να έχουμε περισσότερες συμφωνίες επανεισδοχής και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Όσο λιγότερους ε, παράτυπους μετανάστες έχουμε εδώ στην Ευρώπη, τόσο λιγότερες διαδικασίες επιστροφής θα έχουμε. Η Βουλγαρία που έχει εξωτερικά σύνορα, βάζεται δυνατά της να επιστρέψει όλους όσους έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρώπη. Προσπαθούμε επίσης ε, να παράσχουμε βοηθεία σε όσους δικαιούνται προστασία, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε από μόνοι μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία των εξωτερικών συνόρων με την Τουρκία. Κυρία Γραπίνη, ευχαριστώ. Όπως ε, προκύπτει και από τη συζήτηση, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι στο δημόσιο χώρο δεχόμαστε ε, κριτική ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέχεται κριτική κομισιόν ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ σαφής διάκριση μεταξύ μεταναστών και προσφύγων. Καταρχήν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό δημοσίως και η προσβασιμότητα των κρατών. Σε ό,τι αφορά την υποδοχή προσφύγων ή μεταναστών αυξάνεται, αν οι όροι αυτοί έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια και αν υπάρχουν σαφείς κανόνες, έτσι όπως ε, προκύπτει και από τη σημερινή συζήτηση. Στη συνέχεια, σίγουρα, όπως ε, είπε ο συνάδελφος, εργαστήμαστε ε, για αυτή την οδηγία από το 4 στο 9. Τώρα είμαστε σε άλλο στάδιο. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας και Φυσικά βλέπουμε τι συμβαίνει και όπως έγιναν και στη Σουηδία αυτές οι επιθέσεις. Είμαι πολύ περίεργη να δούμε ποιο είναι το ανανεωμένο σχέδιο δράσης μας, σε τι διαφέρει, ποια πρόσθετα μέτρα παρουσιάζει η Κομισιόν για να έχουμε αφενός σαφείς κανόνες να διαφοροποιούμε τους μετανάστες από τους πρόσφυγες, κανόνες υποδοχής, κανόνες παροχής ασύλου, κανόνες επιστροφής και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένω κάποιες διευκρινήσεις γιατί διαφορετικά δεν είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν με ομοιόμορφο τρόπο και μπορεί να εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα να μην ξέρουν τα κράτη τι να κάνουν με τους ανθρώπους αυτούς. Ε, δεν υπάρχουν ακόμη διμερείς συμφωνίες που να έχουν υπογραφεί με τρίτες χώρες, ε, δεν έχουμε ευρωπαϊκές συμφωνίες όπως είπε η Birgit. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν είναι σαφή κατά την άποψή μου και νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να μας παρουσιάσει ακριβείς διαδικασίες και να τις κοινοποιήσει και καλά έτσι ώστε να καταλάβει και εκείνη η γνώμη τι ακριβώς θέλουμε εμείς με αυτή την πολιτική επιστροφών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κιάνγκη, παρακαλώ. E, um, Θέλω να ζητήσω μια διευκρίνηση σε σχέση με το δικαίωμα του ανθρώπου για την νόμιμη πρόσβαση. Σε πολλά κράτη-μέλη ε, μειώνονται οι προσφυγές στη διαδικασία ασύλου. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ενισχυτικό, γιατί και αυτό συμβαίνει για να έχουμε απλούστευση και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ε, για να γίνει πιο γρήγορα η επιστροφή, ο επαναπατρισμός. Εγώ έχω μια αμφιβολία που είναι η εξή. Δηλαδή, για να κάνουμε πιο γρήγορε επιστροφές ε, τελικά μπορεί να παραβιάζουμε τα δικαιώματα και τη νομική πρόσβαση και δημιουργούμε πολίτε δύο κατηγοριών, Α και Β. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν για να προστατεύσει τα δικαιώματα των ετούντων ασύλων σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ από την αρχή. Είχαμε συνάντηση σκιωδών ε, για έναν από του φακέλου τη Λίμπε. Με βάση αυτά που είπε ο Ντία Δεμέρα, και οι αναμνήσεις που είχε από τότε που πέρασε αυτός ο φάκελος στο κοινοβούλιο, αυτά μου οδήγησαν στο να μιλήσω. Εγώ είχα καταλάβει ότι είχαμε ένα πλαίσιο 18 μήνων κράτησης υπό εξαιρετικές περιστάσεις. Πόσο συχνά όμως τα κρατη θεωρούν ότι υπάρχουν αυτές οι ε, εξαιρετικές ε, περιστάσεις για να παρατείνουν το χρόνο ε, των μεταναστών σε αυτή τη διοικητική κράτηση. Τώρα αλλάζει ο όρος από γλώσσα σε γλώσσα, αν είναι detention ή retention. Μετά είχαμε πληροφορίες όχι μόνο για το μέσο όρο ε, του χρόνου κράτησης ε, των μεταναστών, αλλά και την ε, τιμή που είναι πραγματικά η πιο συχνή και πώς το μετρούν αυτά τα κράτη-μέλη. Γιατί από αποστολές κατά το παρελθόν έχουμε δει ότι τουλάχιστον ένα κράτος μέλος αυτή τη στιγμή, αν όχι παραπάνω, κάθε φορά που μετακινείται ένα άτομο από ένα κέντρο κράτηση σε άλλο, ε, μηδενίζουν ουσιαστικά ε, το ρολόι. Οπότε δεν έχουμε συνολικά τον χρόνο κράτηση. Λέμε 15 μέρε εδώ, 25 εκεί, 30 παραπέρα, χωρίς να έχουμε δηλαδή τον συνολικό αριθμό ημερών κράτηση. Θα ήθελα επίση να μάθω αν τα κράτη-μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη διαδικασιών για αυτούς που θα γίνουν σύντομα απάτριδες ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χώρα η χωρα προελευση τους. Ξέρουμε ότι αυτό είναι θέμα. Μία-δύο χώρε έχουν αναπτύξει διαδικασίε προ αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό γίνεται συστηματικά. Και μετά για αυτούς που δεν μπορούν να επιστραφούν. Ε, είναι θέμα ε, μία επαναπροώθηση ή επειδή ε, η χώρα προέλευσή του δεν του παίρνει πίσω. Πώς θα αναπτύξουμε λοιπόν κάποια πολιτική για να ε, διαχειριστούμε και αυτές τις περιπτώσεις και να μην τους αφήσουμε σε καθεστώς ε, ανέχειας και παρατυπίας για όλες τις προεκτάσεις που αυτό έχει για το άτομο αλλά και για τα κράτη-μέλη. Το Κοινοβούλιο εκπώνησε μία μελέτη ε, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα για αυτό το ζήτημα. Αν δεν έχουμε άλλες πληροφορίες θα πρέπει να την ξαναδούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Παρασκευή που μας πέρασε ένα τρομοκράτη σκότωσε τέσσερα άτομα και τραυμάτισε πολλούς άλλους. Παρά το ότι δεν είχε δικαίωμα να παραμείνει στη χώρα, κατάφερε να κάνει αυτή την επίθεση. Γιατί ήταν ακόμα στη χώρα. Ε, βλέπουμε αρκετούς πολιτικούς ε, και ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν ε, επινοήσει έναν όρο ε, μετανάστες χωρίς χαρτιά κτλ. Μοιάζει με κάποιον καημένο δηλαδή που κάπου έχασε τα χαρτιά του. Στην πραγματικότητα εννοούμε ότι δεν έχει ασχοληθεί καν, δεν ζήτησε άσυλο ή ζήτησε και απορριφκέτησε. Οπότε παραμένουν παρανόμως σε μια χώρα. Δεν ε, έχω... Εγώ δεν το βρίσκω σωστό να αποφασίζει ο καθένας που θα μείνει μόνος του κατά παράβαση της νομοθεσίας. Προφανώς άλλοι πολιτικοί το δέχονται. Το 2013 ε, νυν υπουργό Δικαιοσύνης μας έκανε πλακίτσες ε, για την αστυνομία που έψαχνε άτομα που ε, μένουν παραμένουν στη Σουηδία και λέει μα δεν έχει άλλες δουλειές η αστυνομία να κάνει. Δηλαδή ε, ο κύριος Γιώργενσον θεωρεί ότι δεν είναι δουλειά της αστυνομίας αυτής. Η κυρία Βίξτρομ είχε πει το 2014 ότι αντί να επενδύουμε σε επιστροφές ατόμων που δεν είναι καταγεγραμμένα θα πρέπει να ενισχύσουμε την νόμιμη μετανάστευση. Οπότε η λύση που προτείνει δεν είναι να αναζητούμε αυτά τα άτομα και επιπλέον να αυξηθεί η μετανάστευση στην Ευρώπη. Ως ε, Σουηδί πολιτικός δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν εμπιστεύομαι τη Σεσίλια Βίξτρομ. Αυτοί που μας προειδοποιούσαν για αυτά τα πράγματα και ήθελαν να τα προλάβουν θεωρούμε ότι πρέπει να αντικατασταθεί από εισηγήτρια για την πιο ριζική αλλαγή του συστήματος μετανάστευσης συλλογής. Έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Ο πρόεδρος. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνετε άμεσες επιθέσεις. Ε, ε, είναι σημαντικό, λέει η κυρία Βίνμπεκ. Τέλος πάντων, τελειώστε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτοί των οποίων οι αιτήσει απορρίφθηκαν πρέπει να φεύγουν αμέσως από την χώρα. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να μπορούμε να κρατούμε τα άτομα αυτά μέχρι να επιστραφούν. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι, ε, από τις πρώτες προτεραιότητες πρέπει να είναι η επιστροφή ατόμων. Η κυρία Βίξτρομ μια που με ανέφερε η συνάδελφος ε, και συμπατριώτης μου να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα ε, είναι περίεργο το να χρησιμοποιηθεί αυτή η ευκαιρία για να κατονομάζουμε συναδέλφους ε, στο πλαίσιο των τρομερών επιθέσεων που είχαμε στην Σουηδία με θύματα νεκρούς αλλά σας πω ότι στη Σουηδία αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε μαζί από κοινού ότι το μίσος ε, δεν θα νικηθεί με περισσότερο μίσος. Ότι ο καλύτερος τρόπος να ξεπεράσουμε την τραγωδία, να την ξεπεράσουμε από κοινού και ότι το φως και η αγάπη είναι πολύ πιο δυνατά από την τρομοκρατία και το μίσος. Και θεωρώ ότι ε, αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου σε αυτή την Επιτροπή ο καθένας από μας. Να υπενθυμίσω στη συνάδελφο και σε όλους τους άλλους ότι εκφράσαμε την πολιτική μας βούληση εδώ μέσα. Να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση και 75% του Κοινοβουλίου επεσήμανε την αναγκαιότητα ε, αυτού για το οποίο τώρα μου επιτίθενται. Δηλαδή να υπάρχουν ε, νόμιμες δίωδοι για όσους αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Και αυτό έχει σχέση με την ασφάλεια. Ακριβώς για να ξέρουμε ποιος έρχεται, από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Σε μια χαοτική κατάσταση ε, που κατέρευσε ή μάλλον δεν είχε λειτουργήσει ποτέ το σύστημα ασύλου, δεν τα ξέρουμε αυτά. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει λοιπόν να παραδοθούμε, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή για ε, να είμαστε ενωμένοι και πεπισμένοι ότι η αγάπη, η φιλία, το ευρωπαϊκό πνεύμα θα επικρατήσουν. Ε, επί των όσων ζήσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε στη Σουηδία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την πολύ καλή έκθεση του νέου σχεδίου δράσεις για μια νέα αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, αλλά παραμένουν ανοιχτά κάποια ζητήματα γιατί μιλάμε για 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν το 2017 για τις εθελοντικές επιστροφές, αν κατάλαβα καλά. Και άρα τίθεται το ερώτημα, είναι ευρωπαϊκά κονδύλια αυτά αποκλειστικά. Συνυπολογίζεται εδώ και τα κονδύλια που έδωσαν τα κράτη-μέλη ή υπάρχουν και άλλα ε, προγράμματα των κρατών μελών. Μετά αναρωτιέται κανεί. όταν λέμε ότι μέχρι στιγμής ε, λίγοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία ή επέστρεψαν εθελοντικά, ε, γιατί πόσα μιλάμε. και το ποσό αυτό είναι το ίδιο πανευρωπαϊκά ή αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν εθελοντικά από την Ελλάδα λαμβάνουν άλλο ποσό ε, από αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν εθελοντικά από τη Σουηδία. Ή υπάρχει κάποιος μέσος όρος που συμβουλεύει η Κομισιόν στο σχέδιο δράσης. Οπότε ε, πώς έχει το σύστημα μετά, πώς λειτουργεί, του δίνουμε μετρητά, του δίνουμε με επιταγή και τέλος πώς θα αποκλείσει η Κομισιόν το άτομο αυτό, αν υπάρχουν μέτρητά, να πάρει τα μέτρητά και μετά από έξι μήνες ε, να καταθέσει έτσι σε άλλη χώρα. Μετά δικαιούται και από εκεί ε, λεφτά ή κάποιος, ε, κάποιο μέλος οικογένειας του ιδίου ατόμου. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε. Μίλησαν όλοι, ήθελε κάποιος άλλος να μιλήσει. Κύριε Βερζιά, παρακαλώ. δίσταζα να ζητήσω το λόγο γιατί έχασα την αρχή της συζήτηση. Ήμουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, για την ψηφοφορία για την αναδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου. Έτσι λοιπόν δύσκολα τα παρακολουθούμε όλα αυτή τη στιγμή. Θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις ε, γιατί νομίζω ότι υπόθηκαν κάποια πράγματα στα οποία πρέπει να αντιδράσουμε. Θέλω καταρχήν ε, να δηλώσω την ε, αλληλεγγύη μου στην ε, κυρία Βίξτρομ και στο σύνολο των Σουηδών σε σχέση με τις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις που χτύπησαν τη χώρα της. Πιστεύω ότι ε, κάποιες προσωπικές επιθέσεις εδώ δεν είναι έντιμες και θα σταματήσω εδώ. Θεωρώ ότι είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να εργαζόμαστε και να σκεφτόμαστε αυτά τα ζητήματα. Γιατί όλο ένα και περισσότερο βρισκόμαστε σε μια σχιζοφρενική κατάσταση. Αφενός, Έχουμε την πλειονότητα των βουλευτών που ζητούν περισσότερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν και από την άλλη ένα συμβούλιο των κρατών μελών που θέλει όλο και λιγότερα θέλουν ε, να μην ανακατευόμαστε στις υποθέσεις τους, για να το πω έτσι. Όσο δεν θα έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική που να επιτρέπει ακριβώς ε, να μεταχειριζόμαστε με τον ε, ίδιο αμοιόμορφο τρόπο του σωτούντας ασύλου, με τα ίδια κριτήρια, θα είμαστε σε θέσεις που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε σε σχέση με το σεβασμό του δικαίου γενικά. Όταν ε, βλέπω ότι τα ανατολικά σύνορα ουσιαστικά έχουν γίνει σημεία διέλευση ε, για κάποιου, ενώ τα νότια σύνορα είναι ένα και πιο μπλοκαρισμένα, ενώ η πιο δύσκολη κατάσταση για τις εμπόλεμες ζώνες της διώξης ακριβώς είναι στα νότια σύνορα, αναρωτιέμαι τι ψάχνουμε να κάνουμε εδώ. Μας κρούν τον και κινδύνου οι ΜΚΟ, μας λένε να επαγρεπνούμε περισσότερα για τις συμφωνίες επανεισδοχής και ακόμα όταν γίνονται από τα κράτη-μέλη, επαγρυπνούμε περισσότερο για τους ανθρώπους όπου στέλνονται σε κράτη, όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ελάχιστα δικαιώματά τους. Το κράτη-μέλη στέλνουν πίσω ένα και περισσότερους ανθρώπους. Ε, το είδαμε και με την Τουρκία, με το Αφγανιστάν. Βλέπουμε τι γίνεται με τις χώρες του κέρατος της Αφρικής. Εγώ είμαι και αυτή τη στιγμή αγωνίζομαι για να μην σταλούν πίσω στο Σουδάν κάποιοι Σουδανοί ενώ προέρχονται από τον Ταρφούρ ή από άλλες περιοχές του Νότου. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η ανακοίνωση που μας παρουσιάστηκε μειώνει τελικά τη δυνατότητα των εκούσιων επιστροφών αλλά θέλει με κάθε κόστος να μειώσει τον αριθμό των ετούντων ασύλου και να ε, αυξήσει τον αριθμό των αναγκαστικών επιστροφών. Αυτό δεν μπορεί να είναι η λύση αν θέλουμε να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα δικαιώματα των μεταναστών και αν θέλουμε να εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Γενέβης. Νομίζω δυστυχώς ότι απομακρυνόμαστε λένε και περισσότερο από αυτά. Αν μπορώ να επανέλθω στον κύριο Τουντοράκη. Υπήρξαν ε, πάρα πολλές ποιοτικές ε, παρατηρήσεις εδώ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το Κοινοβούλιο και για τη δική μας Επιτροπή και θέλω να σας ζητήσω να επικεντρωθείτε στο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Κομισιόν υπό την οδηγία επιστροφών. Είστε πολύ συγκεκριμένο. Αναφέρθηκαν ε, κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την κράτηση, τα χρονικά όρια κτλ. Μπορείτε να είστε πολύ συγκεκριμένος σε τι ακριβώς μπορούμε και εμείς να επηρεάσουμε και εσείς σε τι μπορείτε να επηρεάσετε. Μπορείτε να είστε όσο δυνατόν πιο συγκεκριμένος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Επαναλήφθηκε και σε διάφορα σχόλια. Σχετιζόταν με τις συμφωνίες επανεσδοχής και με την ε, γενική συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Χωρίς αυτή τη συνεργασία και χωρίς ε, καλές συμφωνίες επανεισδοχής με τις τρίτες χώρες, δεν μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Συμφωνώ 100%. Σε πολλές περιπτώσεις ο Επίτροπος ε, μίλησε για την προσπάθεια της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία από τι τρίτε χώρε κυρίω για τι συμφωνίε επανεισδοχή. και μιλάμε για ευρωπαϊκέ συμφωνίε, όχι διμερεί. Όμω, όπω ε, κάθε διεθνή συμφωνία, χρειάζονται δύο που πρέπει να συνεργαστούν. Μέχρι τώρα έχουμε επίσης 17 εταίρου από τρίτε χώρε να υπογράψουν συμφωνίε επανεισδοχή και αυτέ οι συμφωνίε λειτουργούν καλά. Είχαμε βέβαια και κάποιες δυσκολίες με το Πακιστάν, αλλά ακόμη και αυτή η συμφωνία τώρα λειτουργεί πολύ καλύτερα εδώ και ένα χρόνο. Όμω για τι συμφωνίε που επαναπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα. Προσπαθούμε να ασκήσουμε κάθε πίεση ε, που μπορούμε, κάθε μόχλευση και με ρώτησε κάποιο ναι, ε, αν ασκούμε πίεση, ναι, το κάνουμε, έχουμε μόχλευση και ε, πέρσι, ιδίω για τι πέντε χώρε που περιλαμβάνονται στο σύμφωνο, το λεγόμενο compact, χρησιμοποιούμε διαφορετικούς μηχανισμούς μόχλευσης, ε, όπου μαζί με τις συζητήσει για την επενεσδοχή φέρνουμε και στοιχεία που σχετίζονται με, άλλα, με άλλους τομείς πολιτικής, εμπόριο, θεωρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε το καλό πλαίσιο συνεργασίας για να μπορούμε να υπογράψουμε τις συμφωνίες επενεσδοχής με τις τρίτες χώρες. Τους τελευταίους μήνες, στην προσπάθεια να είμαστε πιο πρακτικοί, υιοθετήσαμε για κάποιες πιο καινοτόμους ε, προσεγγίσεις και όταν ε, είδαμε ότι μια συμφωνία δεν ήταν έτοιμη, μια χώρα να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία, το χάρη με το Αφγανιστάν, βρήκαμε μόνιμους τρόπους ε, επιχειρησιακούς ή άλλες μορφές συνεργασίας που προσπαθούν τουλάχιστον να είναι σαφείς σε σχέση με τους κανόνες και τις δικλείδες ασφαλείας που ισχύουν. Είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα. Όχι. Ελπίζουμε να καταφέρουμε περισσότερα. Έχουμε τρίτε χώρε κυρίω χώρε προέλευση από τη Δυτική Αφρική, με τι οποίε θα θέλαμε να βελτιωθεί η συνεργασία για την επενδυστοχή. Όμω, εντατικά διαπραγματευόμαστε με τι τρίτε χώρε και ελπίζουμε και φέτο, ε, χρησιμοποιώντα ε, την προσέγγιση του πλαισίου εταιρική σχέση, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με τι διαδικασίε ασύλου για το αν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν όλους τους ε, μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους για να αυξήσουν την ταχύτητα ε, των διαδικασιών ασύλου. Παρακολουθούμε συνεχώς πώς εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη την νομοθεσία περί ασύλου και αυτό αποτελεί τμήμα της συνεχούς αξιολόγησης που γίνεται. Είχαμε και άλλε ερωτήσει σε σχέση με την οδηγία επιστροφών και τους κανόνες για την διοικητική κράτηση ή την ε, φυλάκηση. και ερωτήσεις ε, σε σχέση με τα όρια, αν ε, τα τα κράτη-μέλη ή όχι ή ρωτήθηκε πόσα κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εσωτερικό του δίκαιο. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν μεταφέρει στο εσωτερικό του δίκαιο την οδηγία επιστροφών, περί επιστροφών. Τώρα, σε ποιο βαθμό αυτό είναι άλλο ζήτημα. Όπως σας είπα, εδώ και δύο χρόνια Κάνουμε αποστολές αξιολόγησης έγκεν, κυρίως για τις επιστροφές και στη βάση αυτή έχουμε καταρτήσει τη σύστασή μας. Δεν υπάρχει τίποτα στη σύσταση που εθετήσαμε που να είναι θεωρητικό ή να προέρχεται από μια θεωρητική αξιολόγηση που κάναμε για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή. Όλα προέρχονται από πρακτικές παρατηρήσεις και τα πορίσματα που συλλέξαμε ως μέρος ε, της διαδικασίας αξιολόγησης έγκεν. Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρθηκε η οδηγία στο ιστορικό δίκαιο ή ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν τα χρονικά όρια ε, τα κράτη-μέλη σε σχέση με την κράτηση ή τη διοικητική κράτηση είναι αντικείμενο αυτής της αξιολόγησης. Επικύλουν αυτές οι πρακτικές. Δεν βρήκαμε μέχρι τώρα στις αποστολές αξιολόγησης έγκεν επαρκείς ε, λόγους για να ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβάση, αλλά σκεφτόμαστε αυτή τη δυνατότητα στα πλαίσια τις δυνατότητες αντίδρασης που έχουμε, ανάλογα και με το πώς θα συνεχιστούν οι αποστολές αξιολόγησης έγκεν, γιατί τώρα είμαστε ουσιαστικά στο ίμιση της διαδικασίας. Υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ προσφύγων και παράτυπων μεταναστών, ρώτησε ε, κάποιο μέλος, ναι, πιστεύουμε ότι είναι. Νομίζουμε ότι υπάρχει σαφής διάκριση στην ομοθεσία μας για τις ε, διαφορετικές μεταχειρήσεις και διαδικασίες που εφαρμόζονται στους πρόσφυγες όσου ζητάνε διεθνή προστασία και σε όσους είναι σε παράτυπη κατάσταση και για τους οποίους πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες περί επιστροφής. Νομικές οδοί έναντι αποτελεσματικών επιστροφών. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει τάση να προσθέτουμε να προσφέρουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Είναι τμήμα αυτό που είπα στην αρχή, προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μια δράση στο εσωτερικό του συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης. Κονδύλια για τις πολιτικές επιστροφής και τις διαδικασίες, ανέφερε ο βουλευτής 20 εκατομμύρια. Να αναφέρω ότι σήμερα ως ε, μέρος ε, του Ταμείου Ένταξης και Ασύλου 806 ε, εκατομμύρια έχουν δοθεί για να υποστηριχθούν ακριβώς αυτές οι δραστηριότητες. Το 2017 η Κομισιόν θα δώσει επιπλέον 200 εκατομμύρια για να αυξήσει την ικανότητα των κρατών μελών για τις επιστροφές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχουν τα κονδύλια ε, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οι αρχές των κρατών μελών για προγράμματα και για τις εκούσιες επιστροφές αλλά και για τις αναγκαστικές επιστροφές όπου χρειαστεί. Κάνουμε τη σωστή παρακολούθηση για τις ακούσεις επιστροφές. Εμείς στο EVRR έχουμε συμπεριλάβει και τη συνιστόσα της επανένταξης. Γι' αυτό μιλάμε ε, ουσιαστικά για πακέτα που αφορούν ε, την ε, υποβοηθούμενη ακουστική επιστροφή αλλά και την επανένταξη. Έχουμε και προγράμματα για τις χώρες όπου η επανένταξη είναι ευαίσθητο θέμα για να δούμε πώς ε, επανεντάσσονται οι άνθρωποι στις κοινότητές τους, να βοηθήσουμε τις κοινότητες να επανεντάξουν τους μετανάστες αυτούς και φυσικά με το μικροπρόθεσμο στόχο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανακάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. Σας ευχαριστώ. Okay, very... Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα σταματήσουμε τη συζήτηση για τα σημεία 6-7. 11 και 10 θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Θα κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα μέχρι τότε. Αν δεν έχετε ακόμα την κάρτα σας, μπορείτε να πάτε να την πάρετε. 11 και 10 λοιπόν, ακριβώς παρακαλώ. Okay, colleagues, we're going to begin. Συνάδελφοι, ξεκινάμε με τις ε, ψηφοφορίες. Είστε έτοιμοι. Ξεκινάμε με το πρώτο ψηφοφορία, σημείο 8, κανόνες για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ντανιέλ Φιγιώτη, εισηγητής. Ξεκινάμε τροπολογία 15 αρχή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Θα ε, σταματήσω γιατί υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που μπαίνουν τώρα στην αίθουσα. Θα, ναι, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει ανοιχτή η ψηφοφορία. Κάποια μέρα κάτι θα γίνει και θα φταίω εγώ βέβαια. Λοιπόν, ψήφισαν όλοι. Ωραία. Πέρασε. Δεκτή. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, το μηχάνημά μου δεν δουλεύει. Υπέρ ψήφισα. Μάλιστα. Ωραία. Δεκτό. Το μηχάνημα της κυρίας Σπινέλη δεν δουλεύει, λοιπόν, υπερψήφισε γιατί ήταν δικιά της η τροπολογία. Δεν αν θέλατε να καταψηφίσετε την τροπολογία σας. Α, αλλάξατε θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Ωραία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 19, αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 και 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αδέκτη. Τροπολογία 21. Μέρος πρώτο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 μέρος δεύτερο. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 2. Αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3. Αρχιτή ψηφοφορία. πέρας ε, δεκτή 4 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται ε, 5 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 23 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. 24 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 25 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 26 αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 28 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 1 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 29 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 2 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Ταπολογία 35 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 7 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 36 μέρες πρώτο η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 36 μέρες δεύτερο η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 37, 38, 39 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Εκτιμώντας απολογία 8 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 9 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεκτή. Δέκα άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Έντεκα άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Δώδεκα άρχεται. Δεκτή. Δεκατρία. άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία. Τελική. Πέρας. Δεκτή με πέντε ψήφους κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια. We now uh, move to the... Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 9 για την ε, στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της Europol. Ο κύριος Δίας Δεμέρα θέλει να πάρει το λόγο. Ο Ιδάλλος μπορούμε να περάσουμε απευθεία στη ψηφοφορία. Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες της κυρίας Σίπελ και της κυρίας Κίντσι και άλλοι από τον κύριο Πέτερσον. Δεχόμαστε και τις τρεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δίας Δεμέρα. Ωραία, συνάδελφοι, α περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 51 ψήφι υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ συνάδελφοι τέλος της ψηφοφορίας και της ε, συνεδρίασης. Και τώρα συντονιστές. Ευχαριστώ. Yes, we have 10 break and... Έχουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα.